Dear Συνάδελφοι, θα έλεγα να ξεκινήσουμε και θα μιλήσω γερμανικά. Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, ελπίζω να προσέλθουν και άλλοι ευρωβουλευτές σε αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση που έχουμε σήμερα. Διότι έχουμε μαζί μας εκπροσώπους από από συμμετέχοντες ε, στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Ολέα. Η ακρόαση μας ε, θα μεταδοθεί και στην ιστοσελίδα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη θα μας παρακολουθήσουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα θα μπορέσουν και να συμμετάσχουν μάλιστα. Και εσείς ως ε, ευρωβουλευτές μπορείτε να συμμετάσχετε στην online συζήτηση που θα γίνει με τη βοήθεια του hashtag EYE2018. Αυτό βεβαίως το απευθύνω και σε όλους τους προσκεκλημένους μας και η συζήτηση που θα γίνει στο διαδίκτυο θα εμφανίζεται και εδώ στην, ε, στις ε, οθόνες μας. Θα μπορείτε να βλέπετε. Όπως γνωρίζετε, από το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο διοργανώνει την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία στο Στρασβούργο. Στη φετινή εκδήλωση συμμετείχαν 9.000 νέοι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά υποδέχτηκα και μια ε, ομάδα νέων ανθρώπων που μου έδωσαν ε, πολύ θετικά σχόλια. Λοιπόν, για να εξασφαλιστεί και μια πολιτική συνέχεια στην εκδήλωση αυτή, το Προεδρείο στις 16 Ιουνίου 2014 αποφάσισε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης για την νεολαία να υποβάλλονται πάντοτε στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Η αντίστοιχη έκθεση λοιπόν έχει διαβιβαστεί στους ευρωβουλευτές το Σεπτέμβριο. Και ο σκοπό τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι να υπάρξει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των νέων Ευρωπαίων αφενός και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφετέρου και προκειμένου να ανταποκριθούμε στο στόχο που έχει η ίδια η εκδήλωση για την νεολαία, να ακουστούν οι απόψεις και οι ιδέες των νέων ανθρώπων εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την τρίτη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, λοιπόν, που έγινε φέτος, έχουμε μαζί μας τρεις συμμετέχοντες που θέλουν να μας μιλήσουν για, τους, ε, για τα όνειρά τους, για τις προσδοκίες τους. Θα μας δώσουν ιδέες, δηλαδή θα είναι οι πάροχοι αν θέλετε των ιδεών και εμείς θα είμαστε οι παραλήπτες των ιδεών. Για τα θέματα έχετε ενημερωθεί, οι ευρωβουλευτές θα λάβουν το λόγο, αφού δώσουμε τον, τον λόγο βεβαίως στους προσκεκλημένους μας, για να τοποθετηθούν και εκείνοι. Σε δύο τμήματα θα γίνει αυτή η συζήτηση. Στο πρώτο τμήμα θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και στο δεύτερο τμήμα θα μιλήσουμε για τους νέους και την πολιτική. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω χρόνο επειδή, θέλω να σα παρουσιάσω τους προσκεκλημένους. Έχουμε την Μαλούσε Σεσίλ Βαντράνεν Γκλίσμαν, τον Μάρτιν Ούσελ και την Καρολίνα Χολόβνια μαζί μας σήμερα εδώ στην Επιτροπή. Και θα ξεκινήσουμε με την Μαλού Βαντράνεν Γκλίσμαν, η οποία και θα μας παρουσιάσει τις ιδέες της για την εταιρική σχέση των σχολείων ε, Ανατολής και Δύσης. Δύο λεπτά, αλλά χωρίς να αγχωθείτε αγαπητοί μου, μπορείτε να πάρετε και λίγο περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Για τις εταιρικέ σχέσεις των σχολείων σε Ανατολή και Δύση θέλω να σας μιλήσω εγώ. Στο πλαίσιο τη παγκοσμιοποίηση και του αναδυόμενου λαϊκισμού είναι σημαντικό η γενιά μου να αναγνωρίσει τη σημασία των δημοκρατικών αξιών ω ραχοκοκαλιά τη κοινωνία μα. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνω να υπάρξει ένα πρόγραμμα εταιρική σχέση στον τομέα των κοινωνικών επιστημών μεταξύ σχολείων ε, της, Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την... τα σχολεία την ευκαιρία να συζητήσουν την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προλάβουν το εθνικιστικό περιεχόμενο που συχνά ε, διδάσκεται στις ε, τάξεις μας. Θα χρειαστεί λοιπόν πολλής χρόνος, 50% των, ιστορι... των ε, μαθημάτων ιστορίας και γεωγραφίας από στις τάξεις 9 έως 12 για να διδαχτούν με επάρκεια αυτά τα θέματα. Επίσης, ε, μπορούν να υπάρξουν, ε, αυτή η εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλλει και σε άλλου είδου πολιτιστικές ανταλλαγές. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει ένας πολιτικός διάλογος που θα βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και την εμπιστοσύνη. Οι χώρες που θα αποτελούν τα ζευγάρια θα εναλλάσσονται κάθε χρόνο. Για να υπάρξει βεβαίως αυτή η, αυτή διδασκαλία θα χρειάζεται, να, χρειάζεται βεβαίως ε, ένα συγκρίσιμο επίπεδο γνώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει λοιπόν ένα διαδικτυακό χώρο μελέτης και εργασία με υλικό εκπαιδευτικό αλλά και να χρηματοδοτήσει ταξίδια ανταλλαγή. Επίση, θα πρέπει στη διαδικασία αυτή να συμμετέχουν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονε. Στόχο αυτού του προγράμματο είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να προστατευτούν οι φιλελεύθερε αξίε και να εισαχθούν κοινοί στόχοι εκπαιδευτικοί ω πρώτο βήμα προ τη δημιουργία ενό πανευρωπαϊκού ε, αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης. Ελπίζω λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής σας να ε, πάρουν την ε, δυνατότητα αυτή, αυτή την ευκαιρία ή μάλλον αυτή την ιδέα τη δική μου για να δημιουργήσουν, να πιέσουν ε, στη, προς τη δημιουργία ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος και των αντίστοιχων προτύπων των εκπαιδευτικών που προτείνουν. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε με τον Μάρτιν Ούρσελ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια ιδέα για ε, τα πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μου ιδέα αφορά μια πλατφόρμα πανευρωπαϊκή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φανταστείτε ένα κάμπους, ένα, μια πανεπιστημίου πολύ στην Ευρώπη όπου συγγραφείς, κινηματογραφιστές μπορούν να ζουν, να εργάζονται μαζί και να μοιράζονται τις ιδέες τους με ζωγράφους, ηθοποιούς, παραγωγούς. Φανταστείτε ε, κινηματογραφικά στούδια και τηλεοπτικά στούδιο να συνεργάζονται προκειμένου να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή κοινότητα ε, ανθρώπων που απασχολούνται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φανταστείτε ένα δημόσιο κανάλι τηλεόρασης ε, πανευρωπαϊκό που θα έχει την, ε, ως μοντέλο του το BBC και το Netflix με περιεχόμενο που θα το δημιουργούν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες και που θα παρουσιάζεται στα άλλα μέλη της κοινότητας, όπου θα γίνεται συζήτηση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί η Disney Pixner, έτσι ακριβώς δημιουργεί ε, το, λειτουργεί το HBO και το Netflix. Δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δημιουργών και τους δίνουν και τον έλεγχο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο δημόσιας τηλεόρασης μπορεί να ανταποκριθεί και να αντιστοιχηθεί σε αυτές τις αρχές. Φανταστείτε ένα πανευρωπαϊκό δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι στο ίντερνετ, αλλά και στους κινηματογράφους που θα δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς ε, να δημιουργούν περιεχόμενο, να εργάζονται, να συνεργάζονται, να συνδέουν ε, την τέχνη τους με το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φαντάστε, φανταστείτε τοπικές κοινότητες ε, συγγραφέων, δημοσιογράφων, δημιουργών, σκηνοθετών να λαμβάνουν βοήθεια από αυτό το κανάλι προκειμένου να δημιουργούν τα τοπικά παρακλάδια αυτού του καναλιού. Ε, μαθητείες αλλά και ευθύνη γιατί για να μπορεί να δημιουργηθεί υψηλού επίπεδου ε, περιεχόμενο χρειάζεται να εκπαιδεύσεις κόσμο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο. Αλλά δυστυχώ οι πόροι δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε, θεωρούμε, ένα ευρωπαϊκό δημόσιο κανάλι τηλεόρασης για την εποχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρο. σας ευχαριστώ πολύ για την δεύτερη αυτή ιδέα που προβάλλεται και ερχόμαστε στην τρίτη. Επιστρέφουμε στην ε, Μαλού. Skills at School, δεξιότητες στο σχολείο. Ευχαριστώ πολύ. Τι άραγε θα πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο σε ό,τι αφορά τι δεξιότητε Καινοτομία και δημιουργικότητα είναι τα δύο πράγματα που μπορούν να κάνουν μια κοινότητα να μεγαλώσει. Και τα δύο όμω δεν τροφοδοτούνται αρκετά στα σχολεία σήμερα. Αντί για αυτό έχουν τα παιδιά πολύ περιορισμένη ατομική επιλογή για το τι διδάσκονται και διδάσκονται αφηρημένες έννοιες και τελικώς καταλήγουν να έχουν έλλειψη πρακτικών δεξιοτήτων. Εγώ ως ε, ε, έχοντας συμμετάσχει στο Waldorf σύστημα έμαθα και διάφορα ειδικότερα πράγματα εκτός από τα κλασικά. Από την προσωπική μου εμπειρία μπορώ να πω ότι αυτή η ευρύτερη παιδεία μου έδωσε και την ανεξαρτησία και το θάρρος να αναπτύξω δικές μου ιδέες. Γι' αυτό το λόγο προτείνω ένα αντικείμενο για το σχολείο που να είναι βασισμένο σε project δύο ώρε την εβδομάδα που θα του επιτρέπει στου μαθητέ να μαθαίνουν και διαφορετικά πράγματα. Project-based lessons, μαθήματα project-based, τα οποία θα μπορούν να εφαρμόζονται σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και να λαμβάνουν και πιστοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή του τα παιδιά. Για τέτοια project θα μπορούν να ε, συμμετέχουν και θελοντικά μέντορε. Για παράδειγμα, χειροτεχνικά, ε, οικονομικά, οικιακά από, ε, που να τα μαθαίνουν από ηλικιωμένου ε, πολίτες και, ε, και φωτέρων των φίλων δηλαδή ή τα ψηφιακά ή να μαθαίνουν σχετικά με την πολιτιστική παράδοση των χωρών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου αυτά να μπορέσουν να βρουν μια βάση, ένα πλαίσιο, ένα βασικό εργαλείο, μια βασική εργαλειοθήκη που να μπορεί να παρουσιαστεί μετά από την ολοκλήρωση να μπορούν να βασίζονται σε κριτήρια αξιολόγησης, για παράδειγμα την καινοτομία, που να προσφέρει στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για να αξιολογούνται οι δεξιότητές τους. Για τη μελλοντική αύξηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό θα αποτελέσει την καλύτερη βάση. Για να μπουν αυτά τα μαθήματα project-based στα σχολεία, αυτά θα επιτρέψουν στα παιδιά να αποδείξουν την αξία τους. vielen, vielen. Η πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για τον πρώτο αυτό γύρο παρουσιάσεων των ιδεών σα, Θα ακολουθήσουν τώρα οι ευρωβουλευτέ και πρώτη η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ιδέες. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα του δημοσίου τηλεοπτικού καναλιού. Τι σημαίνει ότι είναι συνδυασμός Netflix και BBC, γιατί το BBC ε, είναι ε, ένα κανάλι συνεχούς ροής, ενώ το HBO και το Netflix ε, βασίζονται στη ζήτηση. Άρα μιλάμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όχι για μια δημόσια τηλεόραση αλλά ψηφιακή πλατφόρμα. Τι σημαίνει επιγραμμική ή μη και τι σημαίνει η συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα γιατί μου ελέγχθη ότι ο δημόσιος τομέας δεν αρκεί. Θα ήθελα να πείτε τη γνώμη σας. σε ευχαριστώ. Σαμπίνε Φερχάιν. Και εγώ θέλω να επανέλθω στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα media. Εδώ θέλουμε να προσελκύσουμε κυρίως, με την ιδέα αυτή, αυτό κατανοώ από την ιδέα δηλαδή, νέους και νέες. Και απευθύνεστε ή στην νεολαία δηλαδή ή σε όλους. Δεύτερο, για την επιγραμμική ή μη, μάλλον για την γραμμική ή μη προσφορά. Διότι μάθαμε ότι για τις νέες γενιές καταναλώνουν λιγότερο γραμμικές ε, εκπομπές, δηλαδή διαρκή ροή, και περισσότερο on demand. Ενδιαφέρει περισσότερο μια Mediatek, μια πλατφόρμα, τι γίνεται επίσης με, τις, ε, με τα προγράμματα ειδήσεων, διότι το Euronews είναι ένας πανευρωπαϊκός σταθμός που βέβαια η εμβέλειά του δεν φαίνεται να ενδιαφέρει πάρα πολύ τους νέους συγκεκριμένα η προσφορά αυτή την οποία εσείς προτείνετε και που θα θέλατε να δείτε πώς θα είναι, τι, τι μορφή θα λάβει. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για το, την καινοτόμα αυτή ματιά στο μέλλον. Καινοτόμα και δημιουργική. Δεύτερο, παρακολουθώ Ακολούθησα έκθαμβη τις ε, δύο παρουσιάσεις των ε, παιδαγωγικών προγραμμάτων, που, των παιδαγωγικών ιδεών που ε, προτείνεται, που είναι σαφής και η ευρωπαϊκή τους θεμελίωση. Είχαμε σήμερα το πρωί τους βραβευμένους με τα βραβεία Καρλομάγνου και αυτό, αυτή η πρότασή σαντάστε νομίζω στην ίδια προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, Λουίτζι Μορνιάνο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο πρώτο θέμα, δηλαδή την εκπαίδευση και τις δημοκρατικές αξίες μέσα από αυτές τις ανταλλαγές Ανατολής ε, Δύσης. Και γιατί κάνω αυτή την παρέμβαση πέρα από όλα τα άλλα γιατί το ερώτημα είναι το εξής. Σήμερα μιλάμε για συνοχή χωρίς αποκλισμούς και για δημοκρατία. Ποιος είναι ο χώρος έμπρακτα του 50% του χρόνου που θα δίνεται για την εμβάθυνση των ε, αξιών. Δηλαδή, επί της ουσίας, ε, ποια είναι τα καθήκοντα και υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα. Νομίζω ότι υπάρχει μία υποβάθμιση των καθηκόντων, αλλά θα ήθελα να ξέρω τη δική σας άποψη. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και το ΆΙ πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ως προς το θέμα των σχολείων και των ανταλλαγών, βεβαίως πρόκειται για ένα πιλωτικό σχέδιο και ανταλλαγές από πρώην ανατολικές χώρες με τη Δύση. Υπάρχει όμως και το Erasmus Συν. Δηλαδή υπάρχει και η βασική δράση 2. Και εδώ μιλάμε και για εταιρικές σχέσεις. Γιατί δεν θα μπορούσατε να υποβάλλετε τέτοια, τέτοια προγράμματα μέσα στα πλαίσια της Key Action 2 του Erasmus Plus, έτσι ώστε να έχετε μία κοινή δράση με τα σχολεία υπάρχει πείρα στον τομέα των, ε, της ευρωπαϊκής, ε, του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Γνωρίζετε λοιπόν ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά σχολεία που είναι πολύ λίγα. Θεωρείτε λοιπόν ότι ίσως θα έπρεπε να διευρυνθούν Δηλαδή η ευρωπαϊκή ηθαγένεια θα πρέπει να προέρχεται από τα κάτω, από τα σχολεία, έτσι ώστε τα σχολεία να μπορέσουν να συμμεριστούν αυτές τις ιδέες. Ως προς την πλατφόρμα, εγώ είμαι η συγγήτρια της Δημιουργικής Ευρώπης. Θεωρείται ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Υπάρχουν ήδη πλατφόρμες μέσα στη Δημιουργική Ευρώπη. Θα μπορούσατε να μας υποδείξετε κάτι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σόφλιν. Δύο λεπτά. Thank you. I very much... Ευχαριστώ. Μου αρέσει πολύ η ιδέα της ανταλλαγής δεξιοτήτων νέων και μεγαλύτερων σε ηλικία. Μ' αρέσει όμως και πολύ αυτή η ιδέα της ε, διασύνδεσης Ανατολής ε, και Δύσης. Ε, Μαλού Σεσίλ, νομίζω ότι είπες κάποια στιγμή ότι πρέπει να προλάβουμε το εθνικιστικό περιεχόμενο για να προστατεύσουμε τις, ε, τις ε, φιλελεύθερες αξίες και τη δημοκρατία. Είναι λίγο οργουελιανό όμως αυτό, διότι κάποιες φορές ε, οι εθνικισμοί έχουν και έναν προοδευτικό χαρακτήρα, γιατί συνδέονται με την προστασία των, των, της πατρίδας, ας πούμε. Αυτό είναι μια γενική άποψη που μπορείς να υποστηρίξεις, γιατί μήπως ε, τελικά καταλήξουμε να θεωρούν άνθρωποι στην Ανατολική Ευρώπη ότι τους πατρονάρει η Δυτική Ευρώπη λέγοντάς τους ότι αυτό που σκέφτονται και αυτό που πιστεύουν δεν είναι σωστό και μήπως με αυτόν τον τρόπο ε, τελικά τους οθήσουμε σε μια πιο ακραία εθνικιστική στάση κάτι που και εσύ από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθείς να, να, αποφύγεις. Ευχαριστώ η κυρία Ζόντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω κι εγώ στην ε, μητρική μου γλώσσα, στα τσεχικά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την δραστηριοποίησή σας, για τις παρουσιάσεις ε, που κάνατε, για τις ιδέες που μας παρουσιάσατε και θέλω να κάνω έκκληση σε εσάς. όσον αφορά αυτές τις σχολικές ανταλλαγές που μας περιγράψατε. Εγώ, από ό,τι κατάλαβα, εμ, ζητάτε μια, ένα καλύτερο συντονισμό, μια τυποποίηση, αν θέλετε, στην, στον τομέα της παιδείας και των αναλυτικών προγραμμάτων στα σχολεία. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος πλούσια. Ταυτόχρονα όμως ε, είναι και μια ήπειρος πολύμορφη. Θέλουμε λοιπόν μια βαθύτερη ε, συνεργασία, αλληλοκατανόηση, αλλά όχι τυποποίηση. Από αυτή την άποψη, θεωρείτε ότι είναι σωστό το αίτημά σας αυτό όσον αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση στην Ευρώπη, στον τομέα και στον, ε, στο θέμα των, της, ε, της ε, ιδιότητας του πολίτη, του Ευρωπαίου πολίτη. Εδώ, εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε συντάξει και έκθεση σχετικά με το αντικείμενο αυτό και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πράγματι να τυποποιηθούν ώστε όλοι οι πολίτε να λαμβάνουν, όλες τις, να λαμβάνουν όλοι τις ίδιες πληροφορίες. Δηλαδή ποιες υποχρεώσεις και ποια δικαιώματα απορρέουν από την ε, ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Λέει, Πρόεδρος, έχω και εγώ μια ερώτηση για το Πανευρωπαϊκό Media Project. Πρόκειται για μια ιδέα η οποία απασχολεί και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν και κάποιες ιδέες από την, ε, το πρώτο γερμανικό κανάλι, το ARD, ένα είδος δηλαδή κλασικής Mediatek. Και αν καταλαβαίνω καλά την πρότασή σας, πρόκειται κάπως για μια ανταλλαγή μεταξύ χρηστών, παραγωγών, καλλιτεχνών. Δηλαδή, να ξεκινήσει μια τέτοια συνεργασία ώστε να προκύψει από αυτήν νέα ενδιαφέρουσα παραγωγή. Αυτά, εάν κατανοήσα καλά. Έχετε την ευκαιρία όμως να τα διευκρινίσετε. Ακόμα τώρα η ε, συνάδελφός μας Julie Ward. Σας ευχαριστώ πρώτα που ήρθατε εδώ στο κοινοβούλιο μας. Κλείνεται έτσι ένα κύκλο. Εγώ δραστηριοποιούμε πολύ ως Ευρωβουλευτής στο European Youth Event και πρόκειται για μια θαυμάσια και πάρα πολύ θετική εμπειρία. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων και στους άλλους ε, ευρωβουλευτές που κατάφεραν να έρθουν εδώ, να παραστούν. Βεβαίω εργαζόμαστε ε, για το όφελος των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τις ε, χώρες μέλη. Είχα μια ομάδα από την βόρειο-δυτική Αγγλία, η οποία με το οποίο ήρθε εδώ, μπόρεσε να έλθει στην Ολομέλεια, στο Εμικύκλο κτλ. Θεώρησε ότι ε, ενδυναμώνεται πολύ. Μπόρεσε να συζητήσει και με ε, ομοτήμους της την Ευρώπη και ε, πολίτες από απομακρυσμένα μέρη της ε, εκλογική μου περιφέρεια, ε, που δεν έχουν και μεγάλε επαφέ ούτε καν μέσα στο Ενωμένο Βασίλειο, είχαν εδώ και έζησαν μια καταπληκτική εμπειρία. Ε, και εγώ ήμουν μία από τα πρόσωπα εκείνα που ε, συνέβαλαν με ιδέε. Άκουσα λοιπόν όλε τι ιδέε που κατέθεσαν οι άνθρωποι αυτοί και τους βρήκα πραγματικά καταπληκτικά επαγγελματίες. Και ξεκίνησε και μια σημαντική πίεση από αυτές τις συνεδρίες ώστε ε, να προωθούν οι ιδέες αυτές ε, και να γίνουν κατανοητές. Πάρα πολύ ωραίο λοιπόν που σας βλέπω εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση Ανατολής-Δύσης, εκεί έχασα λίγο από την εισαγωγή σας. Αναφέρεστε περισσότερο σε Ανατολή-Δύση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός των ορίων. Α, μάλιστα, εσωτερικά, στη, ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει καλώς. Έχω κάποια ε, σχέση και κάποια ευθύνη για τη συνεργασία με τις χώρες της Βαλκανικής. Θα πω λοιπόν ότι οι νέοι τη Βαλκανικής αισθάνονται πάρα πολύ Ευρωπαίοι και δεν θεωρούν αυτούς καθόλου περιθωριοποιημένου. Ε, αισθάνονταν Ευρωπαίοι και πριν ακόμα οι χώρες τους να γίνουν ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω εμπειρία λοιπόν τέτοιου όταν συναντώ με και στι αποστολέ που κάνω στι χώρε αυτέ. Δεν αισθάνομαι καθόλου οι άνθρωποι αυτοί να αισθάνονται λιγότερο ικανοί να ε, ορθώσουν το ανάστημά του και να προβάλλουν ε, το πολιτικό του παράδειγμα και την πολιτική του παρά, ε, παράδοση. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Τώρα θα αναλάβετε και οι δυο το δυσχερέ καθήκον μέσα σε δύο λεπτά να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλε αυτέ τι ερωτήσει. Πολλέ ερωτήσει, σχόλια που δεχτήκατε από διάφορε πλευρέ. Αλλά σα ε, υπόσχομαι ότι θα είμαι γενναιόδορη με τον χρόνο. Ορίστε λοιπόν. Um, Ευχαριστώ πολύ για τις αντιδράσεις αυτές. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν τυποποιημένες ειδήσει για την Ευρώπη, για τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν αφορά τα θεσμικά όργανα, αλλά τις δημοκρατικές αξίες περισσότερο που θα πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία. Δεν μπορώ να πω πώς θα γίνει αυτό, αλλά ένας φίλος μου βρέθηκε στο σχολείο σε μια πρώην ανατολική χώρα, μια φίλη μου, και παρατήρησε ότι υπήρχε πολιτική μεροληψία από τους καθηγητές. Και η μεροληψία προερχόταν από το χώρο της δεξιάς περισσότερο. Εγώ εκτιμώ τους ε, καθηγητές ιδιαίτερα όσο αφορά την ε, διδαχή των κοινωνικών επιστημών. Αν επηρεάζονται λοιπόν, αυτό είναι αρνητικό. Δεν λέω ότι οι νέοι δεν έχουν τις ίδιες αξίες στις πρώην χώρες και στη Δύση, αλλά μέσω των ανταλλαγών βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να ταξιδέψει κανείς παντού και θα μπορούσαμε μέσω ε, μαθημάτων, μέσω Skype να προβούμε σε ανταλλαγές αξιών, γιατί οι δημοκρατικές αξίες είναι κάτι το απόλυτο φυσικό. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το Erasmus Συν. Νομίζω ότι αφορά συνεργασία περισσότερο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, όχι, όχι, Νέβη, η κυρία Κώστα. Εν πάση περιπτώσει δεν αφορά όλα τα σχολεία και τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι ιδιωτικά σχολεία, δεν υπάρχουν σε κάθε πόλη, δεν μπορεί να εγγραφεί το κάθε παιδί εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται η διδασκαλία αυτή σε κάθε επίπεδο δημοσίων σχολείων. Τα σχολεία δεν θα πρέπει να μεροληπτούν ε, πολιτικά θα πρέπει να εμένουν στις δημοκρατικές αξίες που, τη που αποτελούν τη βάση τους. Ναι, έχετε το λόγο. Ωραία. Συνεχίστε. Ο διαπολιτισμικός διάλογος αφορά την προστασία των αξιών δεν πρέπει να υπάρχει επιρροή από το κόμμα που κυβερνά. Το πολιτισμικά διαφορετικό είναι θετικό. Η γλώσσα, οι παραδόσεις, τα έθιμα, όλα αυτά θα πρέπει να διδάσκονται. Αλλά ε, στην ε, ε, διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών υπάρχει μια συμμετοχή 50% αυτών των, ε, αυτής της δασκαλίας που αφορά ε, εθνικά θέματα, αλλά φυσικά κανένας δεν, μπορεί, δεν πρέπει και δεν μπορεί να επιβάλλει αρχές σε άλλους. Ευχαριστώ. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε κάτι. Το Εράσμους παλιότερα πράγματι απευθυνόταν αποκλειστικά σε φοιτητές. Το Erasmus Plus είναι σήμερα πια ένα πρόγραμμα που συνενώνει τα πολλά και διάφορα προγράμματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Ανταλλαγές μαθητών, εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολείων, ανταλλαγές ε, διδασκόντων, ε, ασκουμένων, μαθητευομένων παρέχεται υποστήριξη σε οργανώσεις νέων που υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα αυτά τα κάνει το Erasmus Plus. Ομολογώ ότι τα σχολεία δυστυχώς δεν έλαβαν την απαραίτητη προσοχή στο νέο πρόγραμμα Erasmus Plus. Ε, μίλησα για αυτό το θέμα και χθες με εκπροσώπους των εθνικών υπηρεσιών για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στο μέλλον. Όμως, ανταλλαγές μαθητών σχέσεις μεταξύ σχολείων, όλα αυτά εντάσσονται και εμπίπτουν ε, στο πρόγραμμα Erasmus Για να μην υπάρχει παραξήγηση το λέω. Ε, είναι το πρόβλημα που είχαμε κάποτε με το όνομα, με τον τίτλο του προγράμματος. Λέγαμε παλιά ότι το Erasmus ε, πολλοί πράγματι το συνέδεαν στο μυαλό του με του φοιτητέ και τι ανταλλαγέ ε, στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και είχαμε συζητήσει μήπω να χρησιμοποιούσαμε κάποιον άλλο τίτλο για το πρόγραμμα. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, επελέγει το Erasmus Plus, αλλά νομίζω ότι το διευκρινίσαμε τουλάχιστον εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Κύριε Όρσελ, έχετε και εσείς τώρα τα δύο λεπτά σα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, για τις παρατηρήσεις. Θέλω να μιλήσω πρώτα για το ε, ε, ζήτημα σχετικά με το BBC, το Netflix, την γραμμική μετάδοση και να σας εξηγήσω λίγο τι ακριβώς εννοούσα. Πρώτα απ' όλα, αν κοιτάξει κανείς το μοντέλο του BBC, βλέπει ότι ήδη ε, έχει αρχίσει να αποκτά κάποια χαρακτηριστικότητα λιγότερο γραμμικά. Κάτι που αφορά όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Σε λίγα χρόνια από σήμερα θα δούμε ότι η τηλεόραση θα μεταμορφωθεί σταδιακά σε, μια, σε ένα χωνευτήρι διαφόρων μέσων αν θέλετε όπως, όπως ακριβώς η τηλεόραση παίρνει πολλά χαρακτηριστικά από τον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο φαίνεται να τα καταπίνει όλα τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών μέσων αν θέλετε οπότε η σκέψη μου είναι να, να σκεφτούμε με έναν καινοτρόπο, καινοτόμο τρόπο. Να σταματήσουμε ένα δευτερόλεπτο και να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο σε αυτόν τον ρευστό κόσμο, το νέο, το νέο αυτό ρευστό περιβάλλον. Και η προσέγγιση μου είναι να ε, επικεντρωθούμε στα προβλήματα. Δεν έχω την τέλεια λύση προφανώς να σας προσφέρω, όμως η αφετηρία μου είναι αυτή ότι υπάρχουν τόσοι εξαιρετικοί δημιουργοί στην Ευρώπη. Έχουμε τους καλύτερους κινηματογραφιστές, έχουμε τους καλύτερους δημοσιογράφους, διανοητές, συγγραφείς. Όμως βρίσκονται ο καθένας στο δικό του χωραφάκι και δεν ε, συνεργάζονται, δεν έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλον πέρα από τα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Έχω μιλήσει με πολλούς κινηματογραφιστές και μου λένε ακριβώς αυτό, ότι θα ήθελαν να υπάρχει περισσότερη επικοινωνία, ανταλλαγή αλλά χρειάζεται και μια δομή που θα τους δώσει τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Αν υπάρχει ένας γερμανός κινηματογραφιστής που θέλει να εργαστεί στη Γαλλία, για παράδειγμα, ακούω, μου λένε ότι είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό μου προξενεί αρνητική εντύπωση. Άρα, το ερώτημα για μένα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις ανταλλαγές, πώς μπορεί ο ένας να μάθει από τον άλλον, πώς μπορεί να υπάρξει ένα διαμοιρασμός τη αριστεία που υπάρχει, πώ μπορούμε ο ένας λοιπόν να βοηθήσει τον άλλον για να αρθούμε και στο ύψος των περιστάσεων. Κανείς δεν ξέρει βέβαια ποιο θα είναι το μηντιακό τοπίο στα επόμενα χρόνια, αλλά γιατί να μην το συνδιαμορφώσουμε και εμείς. Όσον αφορά αυτό το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι, το ζητούμενο για μένα είναι να υπάρξει ένας διαμερασμός των ιστορικών των ευρωπαϊκών ιστοριών. Φυσικά όλα αυτά θα ξεκινήσουν από τη βάση, από τις τοπικές κοινωνίες, να μπορούν οι άνθρωποι να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, για τις δικές τους ανησυχίες, την καθημερινότητά τους. Και από εκεί και πέρα βεβαίω θα πρέπει όλα αυτά να εξισορροπηθούν, να μπορεί κανείς να δει διαφορε γενέ, γενναίε από διάφορα γεωγραφικά σημεία και νομίζω ότι εδώ έρχεται πραγματικά το, το κεντρικό ερώτημα. Τι είναι οι αξίες, τι είναι οι ευρωπαϊκές αξίες, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους γύρω από τις ευρωπαϊκές αξίες. Πώς θα μπορούσαμε για παράδειγμα στον Χριστό Κισλόφσκι να του δώσουμε την ευκαιρία να, να μιλήσει, ε, που έκανε αυτή την τριλογία για τα τρία χρώματα, προσπάθησε να, να μιλήσει δηλαδή για, για τρεις διαφορετικές οπτικές ενός θέματος. Βεβαίως ο Κισλόφσκι δεν ζει πια σήμερα, αλλά πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε τη, την δυνατότητα αυτή και σε νέους δημιουργούς. Γιατί φαίνεται και έχω την εντύπωση ότι λείπει από τους νέους δημιουργούς αυτή η δυνατότητα, αυτή η οδός. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Ε, για την κυρία Λιμπάτσικα, μπορείς να πεις αυτό που έχεις ε, προγραμματίσει να πεις στον δεύτερο γύρο. Ερχόμαστε στο δεύτερο γύρο λοιπόν, ε, νέοι, νεολαία και πολιτικοί. Αρχίσουμε με την κυρία, ε, με την Καρολίνα Πολόβνια, Χολόβνια συγγνώμη, Active Citizenship. Έχεις το λόγο. Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να προτείνω ένα βραβείο των ε, ενεργών πρέσβεων της κοινωνίας των πολιτών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις κοινωνικές δραστηριότητες σε όλες τις ε, σφαίρες αποσχόλησης των νέων. Στη ζωή μου προ... Ε, ήρθα σε επαφή με πολλούς καθηγητές, ακόμα και από μικρά χωριά, που δημιούργησαν ευρωπαϊκά κλαμπ για φοιτητές και νέους εργαζόμενους, καθώς και ε, οργανώσεις και συμβουλία νεολαίας. Δεν έχουμε όμως τα κατάλληλα μέσα για να τους ευχαριστήσουμε και να συνεχίσουμε αυτή τη δραστηριότητα για ένα καλύτερο μέλλον. Θεωρώ ότι η πολιτιακή πρέσ, πολιτιακή θα οριστούν από τα γραφεία συνδέσμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έχουμε 10 υποψηφίους από κάθε κράτος μέλος και θα πρέπει να υπάρχει βεβαίως και πλήρης υποστήριξη. Ε, θα πρέπει, θα μπορούν να είναι καθηγητές, ε, νέοι εργαζόμενοι, πολιτικοί, μικιό, ακτιβιστές και όλοι οι νέοι που θα συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Άρα θα έχουμε νέους οι οποίοι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να είναι ε, ενεργοί πολίτες και να γίνουν και πρέσβεις. Έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προωθήσει πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές δράσεις, δημιουργώντας μία χαρτογράφηση όλων των υποψηφίων, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για την θαυμάσια αυτή η ιδέα. Και τώρα πάλι ο Μάρτιν Ούρσελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γειτονιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνω πάλι την προσέγγιση ας πούμε με την εξή ερώτηση, ποιο είναι το πρόβλημα προκειμένου. Αυτό που με απασχολεί εδώ είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα κυριότητας ε, της Ένωσης ως πολιτικής δομής από τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση ότι αυτές οι Βρυξέλλες είναι τόσο μακριά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί και ζει κάπου αλλού. Και νομίζω ότι για να αντιταχθεί κανείς σε αυτό θα πρέπει να σκεφτεί πώς είναι δυνατό να οικοδομηθεί μια πιο προσωπική σχέση ανάμεσα στους ε, ανθρώπους που ζουν στις ε, διάφορες ε, τοπικές κοινωνίες και ιδίως παραμεθόριες με την Ένωση. Ένας τρόπος θα ήταν να δημιουργηθεί ο θεσμός ενός είδους γερουσιαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε πόλη και μικρή και στην περιφέρεια που ο ρόλος του θα είναι ε, ε, ε, εξοκομματικός ας πούμε έτσι και θα έχει πιο πολύ την έννοια να ενθαρρύνει μια αντίληψη για τα τοπικά προβλήματα τα οποία μπορούν να επιληθούν με κάποια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευκολύνει τους πολίτες να λαμβάνουν την βοήθεια από την Ένωση που είτε είναι ήδη δυνατή ή που μπορεί να καταστεί δυνατή. Δηλαδή ξεπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια. Οι φυστάμενες ε, εκστρατείες πληροφόρησης που υπάρχουν ήδη ε, είναι πάρα πολύ απρόσωπες ή ξεκινούν μόνο από τις πρωτεύουσε. Έχω μιλήσει με ανθρώπους στην ε, Ανατολική Γερμανία ή στην Αλσατία με καταστηματάρχες με μικρών καταστημάτων ας πούμε και θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ιδέα για τα προβλήματά τους. Συχνά δεν θεωρούν ότι και η προσωπική τους, η καθημερινή τους ζωή δηλαδή, ε, δεν θα εξυπηρετεί το εάν είχε κάποια ευρωπαϊκή διάσταση. Το καλύτερο λοιπόν είναι να υπάρχουν αυτοί ας πούμε οι γερουσιαστές, σένατορς τους λέει οι οποίοι να προέρχονται από την ίδια την πόλη όπου θα δραστηριοποιηθούν και να, να πάνε να εξηγήσουν στον κόσμο ε, τις δομές, την ιστορία, ε, τους γραφειοκρατικούς μοχλούς, ώστε να βοηθήσουν για παράδειγμα τους νέους να μπορέσουν να αναλάβουν δραστηριότητε και αυτούς δηλαδή που ε, δεν γνωρίζουν πώς να μπουν στην πολιτική. Μπορεί να βοηθήσουν λοιπόν τα πρόσωπα αυτά να ακουστεί η φωνή τους. Έτσι ε, θα μπορέσει και η πολιτική να αντιληφθεί τι ακριβώς χρειάζονται και τι επιθυμούν οι νέοι και οι νέες. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει έργο της Επιτροπής Πολιτισμού, διότι αναφέρεται και στην ε, παιδεία και στην ενεργό ιδιότητα του πολίτου και θα έπρεπε να αρχίσει ήδη πριν από τις ευρωεκλογέ η προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ για την ιδέα σας. Ερχόμαστε την τελευταία ε, ιδέα και το λόγο θα λάβει η Καρολίνα Χολόβνια. Μικροχορηγίες για την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να δίνουν μικρές επιχορηγήσεις για να ενισχύονται τοπικές πρωτοβουλίες εν ώψη και των ευρωεκλογών οι νέοι άνθρωποι, ε, τοπικοί ακτιβιστές, άνθρωποι που ασχολούνται με τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για την νεολαία, υπάρχουν και προσφέρουν, αλλά θέλουν και να το, επιδε... να το αποδείξουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν εξαιρετικές ιδέες, αλλά δεν έχουν τη χρηματοδότηση για να τις υλοποιήσουν. Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζονται πολλές γνώσεις και πόροι για να μπορεί κανείς να ζητήσει χρηματοδότηση. Αυτές οι μικροχορηγίες που εγώ προτείνω είναι πολύ μικρό, μικρά ποσά, ακόμη και 100 ευρώ, που θα μπορούσαν όμως να βοηθήσουν και να ενισχύσουν διάφορες πρωτοβουλίες και project, τα οποία θα μπορούσαν να δίνονται σε εθνικό επίπεδο, ε, ακόμη και από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δίνονται σε συγκεκριμένα project νεολαία. Ένα διαγωνισμό, ένα φεστιβάλ ή ένα εργαστήριο που μπορεί να διοργανωθεί. Ή και μια τελείω καινούρια ιδέα που δεν την έχουμε σκεφτεί ακόμα. Τίποτα δεν ενθαρρύνει τους νέους περισσότερο από την ίδια τη δράση και το να δοθούν χρήματα σε, ε, σε άπειρους νέους μπορεί να ακούγεται ε, επικίνδυνο ή περίεργο, όμως μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση αυτοδιαχείρισης και αυτό μόνο καλό μπορεί να ε, φέρει. Από την εμπειρία μου στο Erasmus Plus μπορώ να σας πω ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ε, φοβούνται αυτή την γραφειοκρατία που συνοδεύει τα περισσότερα ε, ευρωπαϊκά προγράμματα και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό και τα micro grants που προτείνω θα είναι τελείως απαλλαγμένα από αυτό. Η ιδέα μου λοιπόν θα ήταν να ε, υπάρχει μια τέτοια διαδικασία η θα είναι προσβάσιμη σε όλους και που θα μπορεί να διευρύνεται δια, διαρκώς. Κάτι που θα πολλαπλασιάσει την, ε, τον αντίκτυπο με πολύ, πολύ μικρό κόστος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την έκτη ιδέα που μόλις μας παρουσιάσατε. Ξεκινάω με την Κριστίνα που ξαναζήτησε το λόγο. Ελπίζω όμως να τοποθετηθείς για αυτό που μόλις ακούσαμε. Όμως. Ευχαριστώ πολύ. Μαλού. Πολύ σωστά εντόπισε τα προβλήματα με του καθηγητέ, με του διδάσκοντε. Θέλω όμω να σε διαβεβαιώσω. Η Επιτροπή μα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εγκρίνει έκθεση για τον εξυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο έχουμε αφιερώσει στους διδάσκοντες. Και την ανάγκη να έχουν επαρκείς δεξιότητες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στο λειτουργήμά τους. Επίσης, αναφερθήκαμε στην ανάγκη διεύρυνσης και ενίσχυσης τη κινητικότητας ε, στο πλαίσιο του Erasmus Plus. Καρολίνα, για τη δική σου ιδέα τώρα. Ο Κονφούκιος έλεγε ότι αν ένας δάσκαλος διδάξει κάτι στον μαθητή του, δεν μπορεί ο ε, μαθητής ποτέ να ξεπληρώσει, όσο πλούσιος κι αν είναι, ε, αυτήν τη χάρη που του έχει κάνει. Δεν είναι τα λεφτά λοιπόν αυτά που κινητοποιούν ε, τους διδάσκοντες. Εσείς οι νέοι άνθρωποι και οι ιδέες σας είναι αυτό που κινητοποιεί τον, ε, τον δάσκαλο. Όχι η αμοιβή, ο μισθός που θα πάρει. Αυτό που θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο θα ήταν να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων μεταξύ των πρέσβεων, των ambassador και βεβαίως να σας συγχαρώ πολύ για αυτή την εξαιρετική ιδέα για τις ε, μικροχορηγίες που μας παρουσίασες. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενα λίγο να ακούσω τη διερμηνία, λέει η Πρόεδρος. Σίλβια Κώστα, δύο λεπτά. Εγώ θα πρότεινα σε όποιους ε, οργανώνουν τις ε, επικοινωνιακές εκστρατείες να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις προτάσεις γιατί είπατε ότι πολλές φορές οι εκστρατείες παραμένουν στις μεγάλες πόλεις και είναι απρόσωπες. Ως προς ότι ε, τους ε, ενεργούς πρέσβεις εμείς έχουμε ένα νέο πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Ιθαγένεια αξίες και δικαιώματα». Θα μπορούσε να ενταχθεί εκεί η πρότασή σας. Δεν είναι και ιδιαίτερα απλή ή θα μπορούσε να προωθηθεί χωρίς να γίνει μια επένδυση τώρα ή οι γερουσιαστές όπως είπατε ή η Ευρώπη της γειτονιάς σας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί Θέλουμε να καταδείξουμε πώς η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει, να υποστηρίξει συγκεκριμένα project ή προγράμματα. Ως προς τις ε, μικροχορηγίες γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα ε, βραβείο του Ευρωπαίου, του Ευρωπαίου πολίτη της χρονιάς ε, επιδόθηκε χτες. Πρόκειται για 40 πολίτες που επιβραβεύονται. Πρόκειται για μια ενεργή κοινότητα της κοινωνίας των πολιτών. Ως προς τις μικροχορηγίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα κονδύλια ανάπτυξης για την καινοτομία, κοινωνική καινοτομία και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο project να έχει και ε, διαπεριφερειακό χαρακτήρα κατά την άποψή σας. Ο κύριος Μαλινόφ. Ευχαριστώ Φυσικά σας συγχαίρουμε και σας συνεχάρισαν πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ που παραμείνατε στην ουσία και τηρήσατε το χρόνο σας, γιατί έχει μεγάλη σημασία για, το, για τις δημοκρατικές συζητήσεις να μιλάτε για δύο λεπτά. Ακούσατε πράγματα που δεν ξέρετε, προγράμματα και τεκμηρίωση. Αν δεν τα ξέρετε, φταίμε εμείς, γιατί εσείς είσαστε ιδιαίτερα ενεργοί και δραστηροί και αυτό δείχνει τις δικές μας ελλείψεις. Φταίμε εμείς που δεν ξέρετε το εύρος του Εράσμους που λειτουργεί στα σχολεία εδώ και πολλά χρόνια. Όταν υπάρχει μία σύμπτωση απόψεων ε, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στη Βουλγαρία υπάρχει ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Δασκάλου της χρονιάς και το κάνουμε αυτό γιατί υπάρχουν επίσημα κριτήρια που αφορούν το έργο του δασκάλου. Και υπάρχει και μία άλλη μεγάλη ομάδα που μπορεί να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο βιβλιοθηκών ε, στη Βουλγαρία, αλλά δυστυχώς πεθαίνουν οι βιβλιοθήκες. Οι ε, βιβλιοθηκονόμοι ε, έχουν πολύ υψηλές δεξιότητες και θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε και εκείνος Πρόκειται για ένα ε, δίκτυο το οποίο ήδη προϋπάρχει και το πρωί συζητήσαμε ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, αυτό, αυτή τη νέα χορηγία για τον ενεργό πολίτη. Ε, βεβαίως είναι υποσυζήτηση, δεν έχει θεσπιστεί ακόμα, γι' αυτό και είναι κάτι που δεν γνωρίζετε. Ευχαριστώ κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ Πέτρα. Επανέρχομαι στην πρόταση, στην πρόταση για την ανάληψη κυριότητας της ευρωπαϊκής ιδέας από τους απλούς πολίτες. Πράγματι αυτό είναι μέγα καθήκον για μας. Υπάρχει αυτή η έλλειψη ε, κυριότητας, δηλαδή ε, ενστερνισμού, ακόμα και αν δεν πρόκειται για απλούς πολίτες. Είναι και το κοινό μας πολιτικό πρόβλημα, εκτός αν είμαστε αντιευρωπαίοι, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα προτείνεται περισσότερες προσωπικές επαφές. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι πρόκειται για ανάγκη εμπλοκή των πολιτών. Είναι ο μόνος τρόπος για να, και εμπλοκή με τους πολίτες για να προσελκυστεί το ενδιαφέρον του. Δεν μου αρέσει η ιδέα του Σένατορ, του Γερουσιαστού. Τους έχουμε και εδώ, του έχουμε και στις Ηνωμένε Πολιτείε, Είναι πεπαλαιωμένη η έννοια. Στην ε, κάτω Σαξονία μα έλεγαν τότε ότι οι μαθητές είναι οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο από αυτή την ιδέα των ε, γερουσιαστών. Διότι έχουμε πολλούς seniors, ε, senior people, όπως εδώ τον Μαρινόφ που είναι και καθηγητής, είναι πολύ καλύτερα να βάλουμε τους μαθητές να παίξουν αυτόν τον Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και εδώ θα μπορούσαμε ίσως να περιλάβουμε σε αυτή την έννοια του πρέσβεως και τους πολλούς εθελοντές αυτούς που πέρασαν από το πρόγραμμα Έρασμος που έχουν ήδη τις ε, γνωριμίες και τις ε, σχέσεις όλοι αυτοί να γίνουν ambassadors για τις ιδέες αυτές και ε, οι ίδιοι αυτά τα οποία έχουν αποκτήσει ήδη οι ίδιοι να τα μεταδώσουν και σε άλλους και να τους εμφυσίσουν την ίδια επιθυμία ε, να προχωρήσουν σε σπουδές εντός Ευρώπης ε, ή να κάνουν πρακτικές ασκήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ούτω καθεξής. Η Ζαμπίνε Φερχάιεν. Και ως βάση για την παροχή πληροφοριών, το έχουμε πει και άλλες φορές, τα Europe Direct Bureaus, τα οποία είναι επιτόπου, όχι μόνο να μην περιοριστούν, αλλά να διευρυνθούν, να μεγαλώσει ο αριθμό του, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την μείωσή του, Το αντίθετο χρειάζεται, ώστε οι νέε και οι νέοι και γενικώ οι ενδιαφερόμενοι για την Ευρώπη να έχουν και ένα συνομιλητή όπου μπορούν να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες. δεν αρκεί καν ο αριθμός των ευρωβουλευτών ώστε να μπορούν να είναι παρόντες παντού. Και τώρα για τις μικροχορηγίες ή μικροεπιχορηγήσεις. Από καιρό λέμε και ιδίω στο πρόγραμμα Europe for Citizens ή το νέο πρόγραμμα αξιών έχουμε πει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις ιδίως όταν πρόκειται για μικρές υποθέσεις ε, προγράμματα συνειδητοποίησης, ε, ανταλλαγές σε πολύ περιορισμένο ε, πλαίσιο θα πρέπει να είναι πολύ πιο εύκολη από την δύσκολη πρόσβαση που έχουμε τώρα σε ε, προγράμματα που συνεπάγονται ε, μια ολόκληρη βαριά γραφειοκρατία και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν μικροποσά τα οποία να μπορούν να δίδονται με εντελώς μη γραφειοκρατικό τρόπο. Απλώς και μόνο αν αποδεικνύεται ο εύλογος χαρακτήρας ενός project. Να γνωρίζουμε βέβαια ότι τα χρήματα θα καταλήξουν να διατεθούν όντω στο συγκεκριμένο έργο. Κάτι πρέπει να γίνει περισσότερο εκεί. Και θα είναι εύκολο να γίνουν πράγματα μετά με πολύ περιορισμένα οικονομικά μέσα. Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο λεπτά όπω και όλοι οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά, κυρία Πρόεδρε σας να ευχαριστήσω κυρίως τους νέους ε, ανθρώπους που ήρθαν εδώ και παρουσίασαν τις ε, εξαιρετικές και καινοτόμες ιδέες τους. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και την αξία που έχει η συμμετοχή της νεολαίας στη δράση. Αυτό ακριβώς είναι και η αξία ε, της διοργάνωσης τέτοιων είδων, τέ, τέτοιου είδους εκδηλώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία ήταν εξαιρετική, ε, είχε μια φοβερή δυναμική και φαίνεται πλέον ότι βγαίνουν και πολύ συγκεκριμένες ιδέες από αυτές τις διαδικασίες. Θέλω να ε, απαντήσω, να σχολιάσω λίγο αυτά τα νέα προγράμματα, γιατί μία από τις, από τις καινοτομίες που έχει προτείνει η Κομισιόν είναι αυτό το σώμα αλληλεγγύης, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πριν από κάποιες μέρες, αλλά και για, την νέα, για το νέο πρόγραμμα Erasmus ε, έχουμε αυτή την έννοια των project. Τα project αλληλεγγύης, ε, στο Σώμα Αλληλεγγύης και στο Εράσμους έχουμε ε, εντάξει αυτά τα project ε, για την νεολαία και θέλουμε μέσα από αυτά τα project να ενθαρρύνουμε τους νέους να προωθούν και να αναδεικνύουν τις νέες τους καινοτόμες τους ιδέες. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα ότι ένας από τους στόχους μας είναι να ενισχυθεί η προβολή των προγραμμάτων. Γιατί πολλέ φορές ακούστηκε και εδώ ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν ήδη δηλαδή, που δεν αξιοποιούνται όμως. Και πολύ συχνά έχουμε δυσκολία ε, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων μας να φτάσουμε σε, σε που πραγματικά απευθυνόμαστε. Αυτό είναι πραγματικά μια πρόκληση αλλά που το έχουμε αναγνωρίσει και που ε, αποτελεί πραγματικά μέλημά μας για να το βελτιώσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Αν μάλιστα τα καταφέρουμε όλα αυτά τα ωραία project και προγράμματα που έχουμε να τα καταστήσουμε πιο προσβάσιμα, να μειώσουμε, να τα απαλλάξουμε από γραφειοκρατία, ε, τότε νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω όμως πρωτού τελειώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, να δώσω δύο λεπτά στην Καρολίνα και στον Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πρώτα εγώ. Όσον αφορά αυτού τους γεριαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλέον γόνιμη προσέγγιση θεωρώ ότι θα ήταν να σκεφτούμε του, τους ε, φραγμούς που αντιμετωπίζει ένας Ευρωπαίος πολίτης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του. Σκεφτείτε για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται τόσο αποσυνδεδεμένη από τους ανθρώπους, από τους πολίτες της. Γιατί την αισθάνονται οι άνθρωποι τόσο απόμακροι γιατί οι λύσεις που δίνονται τελικά δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες. Και αυτό οδηγεί βεβαίως και στο ερώτημα ποιε είναι οι πραγματικές ανάγκες και πώς τις εντοπίζουμε αυτές. Και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στο ερώτημα πώς ένας πολίτης όπως εγώ, θεωρεί ότι τον ακούν και τον βλέπουν οι από πάνω. Εγώ να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι με ακούτε και με βλέπετε. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις και αυτές οι προσκλήσεις ε, είναι πολύ θετικές, αλλά θα πρέπει και να οδηγήσουν σε κάτι. Από τις απαντήσεις λοιπόν, ε, αν θέλουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, α, τις απαντήσεις αυτές δεν πρόκειται να τις βρείτε μέσα από μια διαδικτυακή δημοσκόπηση πρέπει να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και για να γίνει μια σχέση εμπιστοσύνης χρειάζεται διαπροσωπική επαφή, διαζώσεις, πραγματική. Αυτό εννοούσα με την έννοια του γερουσιαστή. Δεν, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η έννοια του πρέσβη ή του γερουσιαστή ως ενός ε, ηγέτη που θα λέει στους άλλους τι θα κάνουν δεν το πολύ σκέφτηκα να σας πω την αλήθεια. Θεώρησα ότι απλά ε, ε, ε, θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος που ακριβώς επειδή δεν θα είναι επαμοιβή θα πρέπει να έχει κάποια άλλα κίνητρα. Είχαμε και μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, αν θα είναι τίτλος ή αν θα είναι θέση εργασίας. Μπορεί κανείς να πάρει τη μία ή την άλλη στάση. Αλλά πάντως για να είναι ελκυστική θα πρέπει να είναι μια θέση η οποία θα επιφέρει, θα έχει κάποια θετική θετικά πράγματα για αυτόν που θα αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο. Ε, θα πρέπει να μπορεί αυτό που θα αναλάβει αυτόν τον τίτλο να μπορεί να πάει στου ανθρώπου και να τους λέει συγκεκριμένα ποια είναι η άποψή σου για αυτό, ε, ποιες είναι οι ιδέε σου, τι δεν σου αρέσει, κάνε μας κριτική για να, να, να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες μας τη δυνατότητα να τοποθετηθούν ανοιχτά, να μπορεί κανείς να αξιοποιήσει την κριτική που ασκείται εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενθαρρύνουμε δηλαδή αυτή την, ε, την κριτική στάση τηρούν πολλοί πολίτες, να την αξιοποιήσουμε ακριβώς για να μάθουμε ποια είναι τα προβλήματα, πού εντοπίζουν οι πολίτες τα προβλήματα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Γιατί ε, αυτό είναι στην ουσία και στον πυρήνα της ε, η αξία της ε, κριτικής. Ευχαριστώ πολύ. Καρολίνα. Θα ήθελα να απαντήσω στα πολωνικά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι βρήκατε ενδιαφέρουσες τις ιδέες μας, τις απολαύσατε και μας δώσατε την ευκαιρία να τις παρουσιάσουμε εδώ. Σε σχέση με την, την πρόταση για τους ενεργούς πρέσβεις, ε, μίλησα για έναν τίτλο περισσότερο, για ένα βραβείο και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε δασκάλους, ακτιβιστές, εθελοντές και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδεχομένως, διότι πολλές φορές βοηθούν τους νέους. Πρόκειται για ένα βραβείο για τους ενεργούς πολίτες υπέρ των νέων ως προς τις ε, μικροεπιδοτήσεις σε αντίθεση με άλλα βραβεία που χορηγούνται για καλές ιδέες οι μικροεπιδοτήσεις θα μπορούσαν να χορηγηθούν πριν από, από την έναρξη ενός project δηλαδή πρώτα θα μπορούσε να λάβει κανείς τα χρήματα και μετά να προωθήσει το σχέδιο αυτό ή το πρόγραμμα αυτό Επίσης ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι δύσκολο να συμμετάσχει κανείς σε διάφορα προγράμματα. Εγώ είμαι ένας, ε, μια απλή πολίτης, αλλά θέλω να ταχθώ υπέρ της Ευρώπης και θα ήθελα η Ευρώπη να με βοηθήσει και να μου δώσει το ελάχιστο να με υποστηρίξει δηλαδή για να αντιμετωπίσω τα θέματά μου. Ήδη από τα 17 μου, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Και φέτος δείξατε ότι αξίζει τον κόπο και ε, το εγχείρημα αυτό όχι μόνο αξίζει τον κόπο αλλά προσφέρει και πολλές ιδέες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την παρουσία σας εδώ και την παρουσίαση των ιδεών σας. Συνεχίστε, θα σας προτρέψω εγώ, συνεχίστε με την ίδια ενέργεια υπέρ της Ευρώπης και υπέρ της συνέχισης της καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ιδέας. σα ευχαριστώ και πάλι πολύ. Χαίρομαι πολύ που έμειναν και τα νεαρά πρόσωπα τα οποία βραβεύτηκαν με το βραβείο Καρλομάγνου και τους οποίους είδαμε σήμερα το πρωί. Χαίρομαι επίσης που βλέπω και άλλα πρόσωπα από αυτά που συμμετέσχουν στην εκδήλωση για την ε, νεολαία. Ελπίζω να μείνετε σε επαφή μαζί μας Έχουμε και διαρκή επαφή με το European Youth Forum και προσπαθούμε να παραμείνουμε σε συνομιλία και μαζί σας. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ και σας εύχομαι καλό υπόλοιπον τη ημέρα σας εδώ στις Βρυξέλλες. Τώρα θα κάνουμε και θα βγάλουμε μάλλον και την λεγόμενη οικογενειακή φωτογραφία με συμμετοχή όλων των Ευρωβουλευτών και με τα τρία πρόσωπα, αν είναι δυνατόν, και με όλες και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέσχουν στο, στην εκδήλωση για την νεολαία. Μια μεγάλη οικογενειακή φωτογραφία. Αν θέλετε εδώ μπροστά λοιπόν. wir weiter. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, μόλις ε, ε, καλμάρουν και λίγο τα πνεύματα από την συγκίνηση. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο σημαντικό νομίζω θέμα της ημερήσιας διάταξής μας, βεβαίως όλα τα θέματα είναι σημαντικά, την εξέταση του σχεδίου έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ε, η είναι η κυρία Σόιντροβα που είναι και παρούσα. Τώρα, προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών είναι η 26η Οκτωβρίου στις 11. Και, ω γνωρίζετε, δεν έχει περάσει και πολύ καιρό από τότε που βαφτίσαμε το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η επίσημη υπογραφή του νομοθετικού κειμένου στο ε, Στρασβούργο, στην αίθουσα της Ολομέλειας. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον και μια ε, νομική βάση για το Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να δούμε βέβαια και πώς θα συνεχιστεί η δραστηριότητά του μετά το έτος 2021. Είπαμε ότι καλό θα είναι αυτό το αποτέλεσμα που προέκυψε από κοπιώδεις ε, συζητήσεις σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή του να το πάρουμε και να κάνουμε copy-paste. Κάτι το οποίο ίσως ε, να διευκολύνει και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιες νέες προτάσεις σχετικά, άλλα τα οποία είχε αρχικά στο κείμενο τα έχει αφαιρέσει, ώστε θα πρέπει παρόλα αυτά να κάνουμε τον κόπο να εξετάσουμε το κείμενο σε βάθος και νομίζω ότι καλά θα κάνουμε όλα όσα έχουμε διαπραγματευτεί να τα περιλάβουμε στο νέο σχέδιο κανονισμού, γιατί δεν χρειάζεται κάθε φορά να εφευρίσκουμε εκ νέου τον τροχό. Νομίζω ότι θα είναι σωστό και σκόπιμο αυτό και εν ώψη των ε, διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο Υπουργών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σόιντροβα για να μπορέσει να παρουσιάσει την εκθεσή της. Ας πούμε πέντε λεπτά. Ναι, μου αρκούν, λέει η κυρία Σόιντροβα. Λυπάμαι διότι οι νέοι αποχώρησαν γιατί τους αφορά άμεσα το ζήτημα. Πρόκειται για υποστήριξη της νεολαίας. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι εισηγήτρια αυτής της πρότασης κανονισμού βασίστηκα στις συζητήσεις προγενέστερων κανονισμών αλλά και μία συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και την Επιτροπή. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα από την ε, τρέχουσα διαδικασία Αυτό που έχει σημασία είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της κοινωνίας και οι ε, εθελοντές και οι συμμετέχοντες να μπορούν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Προτείνω λύσεις στα πιο προβληματικά ζητήματα που καλύψαμε από τις προγενέστερες διαπραγματεύσεις για το προηγούμενο ε, το προηγούμενο σώμα ανηλεγγύης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Helga Truppel στον τριμερή υπήρξαν ορισμένα ζητήματα που δεν ελήφθησαν υπόψη από την πρόταση ιδιαίτερα, ορισμένοι ορισμοί. Επίσης θα ήθελα να υπάρχει μια ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες έτσι ώστε ο εθελοντισμός να είναι η βάση του προγράμματος 86% για εθελοντική εργασία 8% για εργασία και 6% για ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για μία ενδεικτική κατανομή. Το 80% αφορά την εργασία και μαθητεία. Ε, στον τριμερή λάβαμε υπόψη και την ενσωμάτωση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτό το αρχικό 90%. Το Σώμα Αλληλεγγύης δεν αντικαθιστά τα εθνικά προγράμματα. Θεωρώ ότι σε χώρες που υπάρχουν λιγότερες δραστηριότητες η μόνη λύση είναι ο εθελοντισμός. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τη συμμετοχή των χωρών ανάλογα με τον απότερο στόχο. Πρότεινα και άλλες αλλαγές. Θα ήθελα να ενισχύσω το ρόλο των εμπλεκομένων φορέων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να εγκριθεί ως κατεξουδιώτηση πράξη και όχι εκτελεστική. Θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη ορατότητα του σώματος. Η πρόταση της Επιτροπής είναι φιλόδοξη και μιλά για μεταξύ 3 και 50 χιλιάδες Φτάνουμε δηλαδή συνολικά στις 350.000 διορθώνει η ομιλήτρια και γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε και στους εθελοντές. Θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η εργασία χρησιμοποιώντας και τα ΜΜΕ. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη δραστηριότητα και στις απομακρυσμένες περιοχές θα πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο των πρέσβεων και θα πρέπει να συμμετέχουν και σε δραστηριότητες εκπαίδευσης. Η πρόταση τονίζει την ένταξη, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη στοχοθέτηση, δηλαδή αυτοί που έχουν ε, λιγότερες δυνατότητες θα πρέπει να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με μερική απασχόληση. Επίσης θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των στόχων του προγράμματος. Είπα ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς και μας ενδιαφέρει βεβαίως και οι ενδιαφέρουν και οι δραστηριότητες ανατύπω για εργασία και μαθητεία και για τις ανθρωπιστικές ε, δραστηριότητες. Επίσης, για τον εθελοντισμό θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε και τον ορισμό της αλληλεγγύης, γιατί και ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη είναι ύψης της σημασίας. Επίσης, η ΔΕΒ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην ανθρωπιστική διάσταση του σώματος. Ε, εγώ προέβη στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων και η Επιτροπή Απασχόληση συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Αναμένω λοιπόν τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστούμε. Αν δεν έχει αντίρρηση κάποιος άλλος σκιώδης, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαρή Τερέζ που άντεξε μέχρι εδώ παρόλο που είναι άρρωστη. Θέλει όμως να, συνεχίσει, να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό και της δίνω το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μικαέλα Σόντροβα για την εξαιρετική εργασία αυτού του προσχεδίου. Επίσης, την καρποφόρα συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες και υποδείξεις του νέου κανονισμού. Οι διαπραγματεύσεις του προηγούμενου δεν ήταν εύκολες και είναι δύσκολο να μπουν σε ένα νέο αυλάκι μέσω του νέου ΠΔΠ. Συμφωνώ με πολλές τροπολογίες το κείμενο της Επιτροπής και τη μεγαλύτερη ορατότητα και ορίζοντα αυτού του προγράμματος μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας προς τους νέους. Κρίμα που έφυγαν από τη συνεδρίαση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχική δραστηριότητα διαβίου εθελοντισμού. Δηλαδή, ο εθελοντισμός δεν θα πρέπει να είναι στιγμιαίος, αλλά να μετατραπεί σε τρόπο ζωής. Επίσης, θα πρέπει να μιλήσουμε για μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Έχει μεγάλη σημασία ποιες οργα... οργανώσεις συμμετέχουν, αν είναι κοιό ή όχι και ούτω καθεξής και κατά πόσο μπορεί να υπάρχει εθελοντισμός και στην εργασία. Θεωρώ ότι η εργασία θα πρέπει να μην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και θα πρέπει να βασιστούμε στην ποιότητα των δραστηριοτήτων. Θα ήθελα να θυμηθεί η συγγήτρια ότι η αλληλεγγύη είναι ύψης της ε, σημασίας για το κοινό καλό και γι' αυτό θα πρέπει να συνδράμουμε και μέσω αλληλεγγύης και μέσω εθελοντισμού συμφωνώ για υποστήριξη εκ των προτέρων και ε, εκ των υστέρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη Μικαέλα και είμαι σίγουρη ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά στη σύνταξη αυτού του κανονισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Σίλβια Κώστα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ την εισηγήτρια γιατί συμμετείχαμε και εμείς στην ε, διαδικασία διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και γιατί συμμερίζομαι και τις παρατηρήσεις σου και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το ότι ανακτήσαμε τους ορισμούς. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει επί ε, Τρούπελ. Μιλήσαμε για τους συμμετέχοντες, την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα την ποιότητα. Γιατί εδώ δεν γίνεται μνήα για τον χάρτη καθηκόντων και δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ξαναενσωματωθεί. Συμφωνώ με την κατανομή του προϋπολογισμού την δίκαιη αυτή κατανομή δηλαδή και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για σχέδια που αντικαθιστούν τα εθνικά σχήματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία συνεργατική προσέγγιση. Θεωρώ ότι οι οργανώσεις ε, που συμμετείχαν και συμμετέχουν θα πρέπει να ε, συνεχίσουν την ενεργό δραστηριότητά τους. Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι ύψης της σημασίας, ίσως υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ε, έχει σημασία η συμμετοχή των νέων σε μία χώρα και με νέους από άλλες χώρες ως προς την εξισορρόπηση με το θέμα της απασχόλησης θα πρέπει να δούμε και τα κριτήρια και τον προϋπολογισμό, δηλαδή μιλάμε καταρχήν για εθελοντισμό και θα ήθελα να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα έχει η διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας, πώς θα συνεργαστούν οι γενικές διευθύνσεις καθώς και το ζήτημα των ε, εθνικών κέντρων. Και τέλος, θα πρέπει να κατανοήσουμε κατά πόσο θα υπάρχουν εγγραφές από την ιστοσελίδα. Ε, ο θεωρώ ότι ο ισχύων κανονισμός έχει ε, αποδυναμωθεί. Γίνεται λόγος για ενδυνάμει παρουσίαση σχεδίων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δώσουμε μία συνέχεια, γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε και μία κουλτούρα του εθελοντισμού. Helga Ευχαριστώ. Αυτό που είπε ο νέος ήταν αυτή η έννοια της κυριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό συνδέεται με το πρόγραμμα γιατί μιλούμε εδώ πραγματικά για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων και νομίζω ότι ήρθε πια η ώρα μετά την πρώτη αυτή φάση ε, τώρα πια που έχουμε την νομική βάση να βελτιώσουμε το αυτό της αλληλεγγύης και αυτό είναι δουλειά τη δική σου Μιχαέλα εγώ θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να σε υποστηρίξω σε αυτό όλα αυτά που ανέφερε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά ε, και, και οι άλλοι ομιλητέ, ο εθελοντισμός δηλαδή ως ε, μια στάση ζωής ε, και η συμβολή στο κοινό καλό αν θέλετε γιατί αυτό συνδέεται με αυτή την αίσθηση της κυριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά το σημαντικό ερώτημα πέρα από όλα αυτά που μας ενδιαφέρει πώς θα εμπλέξουμε τους ενδιαφερόμενους είναι το αν θα στεφτεί με επιτυχία ο προπολογισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή η πρόταση τη Κομισιόν είναι να ενισχυθεί ο προπολογισμό. Και όπω πάντοτε, όταν μιλάμε στα για προγράμματα, εξαρτώνται από τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφεί ω Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία και απέναντι σε όλους τους ε, συναδέλφους μας ότι χρειάζομαστε επιτυχία ακριβώς για να δοθεί η αίσθηση στους πολίτες ότι τους ανήκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, είναι το διακύβευμα. Και αυτό είναι για το κοινό καλό, ε, είναι για, το, για την προσωπική ανάπτυξη το να συμμετέχει κανείς σε ένα τέτοιο σώμα αλληλεγγύης και στον εθελοντισμό εν γέννη. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μπίλντ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τον Ιούνιο του 2017 είπα ότι δεν υπάρχουν σαφή γεωγραφικά όρια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν θα ε, επεκτηνόταν και σε τρίτες χώρες, όπως πρότεινε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2018 Είπα ότι δημιουργείται ανθρωπιστικός τουρισμός και τίποτα άλλο. Οι νέοι Ευρωπαίοι θα πούν σε μία τρίτη χώρα καταρχήν για να κάνουν τουρισμό και μετά για ανθρωπιστικούς λόγους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, θα υπάρχει και συμμετοχή και από άλλους φορείς οι οποίοι είναι αμφισβητήσιμοι. Πολλές φορές λοιπόν υπάρχει κακοδιαχείριση χωρίς να το ξέρουμε. Άρα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θεσμοθετείται. Δεν είναι επιτυχές πάντα χωρίς ε, να φτάσουμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων, φτάνεται σε μία έλλειψη επικοινωνίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μία τέτοια κίνηση, γιατί οι φορολογούμενοι της Ευρώπης δεν θα το δέχονταν. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν. Αλλά πρωτού το κάνω θέλω να της απευθύνω και ένα ερώτημα. Υπάρχουν, υπάρχει πείρα πλέον ε, με την υλοποίηση του και την εφαρμογή αυτού του σώματος αλληλεγγύης. Ξέρετε ότι είχαμε πολλές διαφωνίες εδώ στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την κατανομή των, ε, των χρημάτων. Τελικά καταλήξαμε στο 90-10, αν δεν κάνω λάθος, κάτι που ζητήσαμε κι εμείς. Όμως έρχονται πάλι ε, αιτήματα από την Επιτροπή Απασχόλησης για να αλλάξει η αναλογία της χρηματοδότησης και να γίνει 80-20. Ερώτημα προς εσάς λοιπόν. Υπάρχει από πλευρά σας κάποια εμπειρία, έχετε συλλέξει στοιχεία, πού θα βασιστείτε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Πόσοι συμμετέχουν σε αυτήν τη διάσταση του προγράμματος και πόσοι συμμετέχουν στην άλλη διάσταση ε, του προγράμματος. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξέρουμε αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Έχετε το λόγο, αν θέλετε βεβαίως. Ε. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Για την ερώτησή σας, ας έρθω στη δική σας ερώτηση πρώτα. Το Σώμα Λυγγύης, όπως είπατε ειδική εισαγωγικά, εγκρίθηκε στις 4 Οκτωβρίου. Σήμερα είμαστε 10 Οκτωβρίου, άρα έχουμε 6 ημέρες από την αρχή ισχύω της νέας νομικής βάσης. Για την ώρα, θα αντιληφθείτε, δεν υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, που τόσο ή είναι πολύ σύντομο διάστημα μετά από την θέση σε ισχύ. Μπορώ να σας δώσω λοιπόν μόνο ενημέρωση για την πρώτη φάση του European Solidarity Corps που είναι και το αποτέλεσμα διαφόρων προγραμμάτων που έχουν στόχο μια κοινή προσπάθεια βασισμένα στην ίδια ε, βάση. Δεν έχω επισκόπηση όλων των προγραμμάτων, άλλοι συνάδελφοί μου ίσως έχουν. Αλλά η συμβολή του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Σώματος έχουμε περίπου 8.000 θέσεις και για το easy call είναι πολύ χαμηλότερο. 53. Εδώ οφείλω να επιμείνω ότι έγινε με διαφορετικό τρόπο εφαρμογής, δηλαδή ήταν εξειδικευμένη πρόσκληση προσφοράς με συγκεκριμένους εταίρους που εργάζονται με διαφορετικό τρόπο. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως ένδειξη για το πώς θα λειτουργήσει η πτυχή της απασχόλησης διότι εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια μεθοδολογία για την οργάνωση του project και να ζητήσουμε υποβολή προσφορών όπως έχουμε συνηθίσει ε, ε, στον Ευρωπαϊκό Θελοντισμό και για να παρακολουθούμε και το έργο. Αυτά βασίζονται ούτως ή άλλως πολύ στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα Ερασμοσύν. Θα απόσχω λοιπόν από του να λάβω ως παράδειγμα το Easy Call ως benchmark, ως ορόσημο για το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και μπρος το σώμα αλληλεγγύης. Υπενθυμίζω επίσης και χαίρομαι για το feedback ότι είναι καλός ο συμβασμός. Έχουμε κανονισμό τώρα τον οποίο συζητήσαμε δια μακρόν και από την πλευρά της Επιτροπής θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικός ο συμβιβασμός. Και όταν θα κάνουμε την επόμενη πρόταση, η ιδέα μας είναι να παραμείνουμε στο πνεύμα του συμβασμού. Υπάρχουν αλλαγές, όπως θα έχετε δει, που προκύπτουν από διαφορετικούς λόγους. Και πρώτο, διότι υπάρχει ανάγκη να είμαστε συνεπείς με την συνολική παρουσίαση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των υπολείπων κανονισμών. Δεύτερο, χρειάστηκε να κάνουμε αλλαγές εκεί όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι που υπαγόρευσαν τις αλλαγές αυτές για λόγους συνεκτικότητας αλλά και για να μπορέσουν οι νέες προτάσεις να περιλάβουν νεαρούς εθελοντές και από ξεχωριστό πρόγραμμα από το ε, ανθρωπιστικό, δηλαδή την ανθρωπιστική διάσταση. Αυτό που θελήσαμε είναι να υπάρχει μια ενιαία είσοδος για τους νεαρούς εθελοντές σε Solidarity Projects και να μην δημιουργηθούν παράλληλες δομές και συστήματα για την απορρόφηση αυτών των νεαρών εθελοντών. Άλλο ήταν ότι Θελήσαμε να είναι λιτό το κείμενο, χωρίς να φορτωθεί με υπερβολικέ λεπτομέρειες που θα πρέπει να ενταχθούν πια στη φάση της εφαρμογής και όχι στον ίδιο τον κανονισμό. Και βρήκαμε επίσης ότι χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση σχετικά με το ποια πράγματα θα πάνε στην εισαγωγική έκθεση και ποια θα μπουν στο καθαυτό τμήμα του κανονισμού, στα άρθρα και από όψη νομικών διατυπώσεων προσπαθήσαμε να βάλουμε και του όρου υπό του οποίου θα γίνονται, θα γίνονται οι συνεργασίε. και αυτά τα βάζουμε στα άρθρα και τι επεξηγηματικές δηλώσει τι βάζουμε στην εισαγωγική έκθεση. Γι' αυτό το κείμενο του κανονισμού θα σα φανεί λίγο διαφορετικό από τον κανονισμό που μόλι τέθηκε σε ισχύ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε πάντως για να παραμείνουμε μέσα στο πνεύμα του συμβασμού ο οποίος επιτεύχθηκε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Όλες και όλοι, αυτό που θα πρέπει να θέλουμε θα είναι αυτά που συμφωνήσαμε στον τριμήρη διάλογο να ισχύσουν, να μην τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή, να δείτε πού ενδεχομένως χρειάζονται κάποιες προσαρμογές ή βελτιώσεις, αλλά να μην αμφισβητηθεί ολόκληρο το περιεχόμενο του πακέτου εξ αρχής. Η Μικαέλα Σόιτροβα Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και για τα σχόλια. Χαίρομαι διότι συμμεριζόμαστε τους βασικούς στόχους αυτού του κανονισμού και έχουμε την ε, ίδια ε, αντίληψη. Βεβαίως ο προϋπολογισμός είναι ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αναμένω τις τροπολογίες σας και θα έχουμε τη δυνατότητα να τις συζητήσουμε. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους σκιώδεις. Είναι πολύ σημαντικό και για εμένα την ίδια. Όπως είπε η κυρία ε, Μπίλντ, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, άμα θέλετε να συμμετάσχετε στη διαδικασία συνεργασίας, ε, είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μία καλή επικοινωνία, διότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι κάτι πολύ χρήσιμο για τους ανθρώπους. Δεν είναι ε, ένα γραφείο τουρισμού. Σας ευχαριστώ πολύ και προσμένω στη συνεργασία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο από εδώ και πέρα έργο σας, αν και θεωρώ δεδομένο ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Υπενθυμίζω άλλη μια φορά, 26 Οκτωβρίου 11 το πρωί είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ψηφοφορία θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου εδώ στην Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή αρκετό καιρό ακόμη. για να εξευρεθούν και οι αναγκαίοι συμβιβασμοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο συνάδελφος Ζαγοράκης είναι εδώ μαζί μας, γι' αυτό και μπορούμε να περάσουμε απευθείας στο σημείο 14. Θέμα είναι η εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Πρόκειται για την αναδιατύπωση μιας οδηγίας μια οδηγία έλεγα λοιπόν και θέλω απλώς να πω ότι προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 16 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου εδώ στην Επιτροπή. Ο λόγος στον συνάδελφο Ζαγοράκη για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Πέντε λεπτά έχετε κύριε Ζαγοράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη. Είναι στο τέλος, γι' αυτό ίσως υπάρχει μια κουράση κόπωση. Λοιπόν, η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη μέσα από τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας επίσημα κρατικά δεδομένα. Τα ανοιχτά δεδομένα αποτελούν πράγματι έναν εκμετάλλευτο θησαυρό κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη τη οικονομία. Η αναθεώρηση τη οδηγία για τη χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα τον Ιούλιο του 2013 σωστά επέκτηνε το πεδίο εφαρμογή, εντάσσοντα και τα μουσεία και τι βιβλιοθήκε στην υποχρέωση παροχή ανάλογων πληροφοριών. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο από την αρχή και η τωρινή αναδιατύπωση τη οδηγία από πλευρά επιτροπή κινείται προς σωστή κατεύθυνση, καθώ μειώνει τα εμπόδια στην αγορά για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για εμπορικού σκοπού. Βεβαίω αυτό θα πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό και τήρηση των κανόνων που έχουμε σε εφαρμογή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονό ότι η παροχή αυτών των δεδομένων και το άνοιγμα τη αγορά δεν θα επηρεάσει ευαίσθητου τομεί, όπω είναι η ασφάλεια, Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια καλή ισορροπία σε αυτό το πεδίο, χωρίς να γίνουν μεγάλες παραχωρήσεις. Όσον αφορά τα θέματα της Επιτροπής μας, η πρόταση της Κομισιόν να διατηρήσει αμετάβλητη την ισχύουσα αντιμετώπιση των φορέων του πολιτιστικού τομέα, όπως παραδείγματος χάρη βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία, είναι επίσης σωστή, δεδομένου ότι η οδηγία στον τομέα αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά. Στο κομμάτι των δημοσίων επιχειρήσεων θεωρώ ότι οι διαδικασίες που θα προκριθούν θα πρέπει να σέβονται τις αρχές του θεμητού ανταγωνισμού και να μην βρεθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται και λειτουργούν στην ίδια αγορά. Το διοικητικό και οικονομικό κόστος είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Τέλος, η πρόθεση της Επιτροπής να ορίσει μέσω καταξακολούθησης πράξη ορισμένε πράξης ορισμένες βάσεις δεδομένων υψηλή αξίας του δημόσιου τομέα δεν είναι επί της αρχής κακή. Θα πρέπει ωστόσο ο κατάλογος αυτός να είναι όσο το δυνατό πιο σαφής και λεπτομερής, ώστε να διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για όλα όσα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν θέλω να με ακρηγορήσω. Προτιμώ πραγματικά να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Όπω θα έχετε δει και στο κείμενο που κατέθεσα, έχω προτείνει ένα μικρό αριθμό τροπολογιών που έχουν στόχο περισσότερο να διευκρινίσουν ορισμένα σημεία Πιστεύω ότι σε συνεργασία με όλε τι πολιτικέ ομάδε μπορούμε να καταλήξουμε σε ευρύτερε συνενέσει είτε μέσω συμβιβαστικών τροπολογιών είτε μέσω υποστήριξη μεμονωμένων τροπολογιών που θα τύχουν ευρύτερη υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε για την σύντομη και ακριβή τοποθέτηση. Δυστυχώς οι άλλοι ο ηγητές δεν είναι παρόντες με μια εξαίρεση. Α, α εσύ είσαι πάλι. Ωραία. Και η Helga Trüppel λοιπόν. Και θα ακολουθήσει η κυρία Μπίλτ. Δεν είχαμε μάθει ακόμα ότι η Helga Trüppel είναι πια σκιώδης ηγητρία. Είμαι πάντα, εκτός αν υπάρχει εξαίρεση και τότε θα σου το πω. Ευχαριστώ τον εισηγητή Νομίζω ότι η προσέγγισή σας, ε, κύριε συνάδελφε, είναι σοβαρή και μετρημένη, διότι ακολουθείτε την πρόταση και τις γραμμές ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για όλους, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να μην διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής κλπ. Είναι πολύ σαφής ο ορισμός της εκ νέου χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Ελπίζω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες οντότητες να μπορούν να υποφεληθούν, αλλά βέβαια πάντοτε με ορισμένους κανόνες. Δεν ζητούμε αλλαγή των κανόνων, ζητούμε παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες. Κάτι που για μένα γενικώ είναι απολύτως εντάξει. Εξέτασα και τις τροπολογίες, σας έριξε μια πρώτη ματιά λοιπόν. Συμφωνώ απολύτως, μετά από μια πρώτη ανάγνωση είναι σαφές για μένα ότι κάνετε του ορισμού ακόμα πιο ξεκάθαρους και ότι αναζητείτε μια καθαρή προσέγγιση για την χρήση και αυτή η κάτοχη των, πληροφοριών του δημόσιου τομέα δεν είναι κύριοι, δεν είναι αποκλειστική κυριότητά τους. Είναι λοιπόν ε, λογικά αυτά που προτείνεται. Θα τις ξανακοιτάξω τις ε, τροπολογίες, αλλά έως τώρα βρίσκομαι απολύτω πάνω στη γραμμή που προτείνεται. Ευχαριστώ, Χέλγκα Η κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ισηγητά η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα δεν αποτελούν βιακή βεύμα στη Γαλλία γιατί είμαστε η τέταρτη ε, χώρα στον κόσμο για την ψηφιακή διαχείριση. Αυτή η κατάταξη έγινε από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει όμως να πω ότι όταν η Επιτροπή μιλά για, για τον ανώνυμο χαρακτήρα των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη γιατί η επαναταυτοποίηση πολιτών σε ομαδοποίηση έχει προχωρήσει και η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί, δεν μπορεί πια να αντιμετωπίσει το θέμα. Μία μελέτη του MIT το 17 μιλούσε για τις τραπεζικές συναλλαγές και ε, σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτότητας και γι' αυτό ε, στη συνέχεια μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση αλλά μόνο για το 90% των πολιτών. Ε, ως προς τροπολογίες οι δικές μου δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη έτσι κι αλλιώς και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προχωρήσει το θέμα από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ζαμπίνε Φερχάιν. Μια σύντομη παρατήρηση από πλευρά μου. Είμαι ε, σκιώδης στην Επιτροπή Εσωτερική αγορά, Αύριο θα έχουμε ψηφοφορία και εξ όσων έχω δει και ακούσει ε, και εκεί κινούμαστε στην παρόμοια, σε παρόμοια κατεύθυνση. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ε, τους πολιτικούς οργανισμούς με ανετιολόγητο τρόπο. Απλώς ε, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πώ τα, τα δημόσια δεδομένα, που έτσι και είναι δημόσια δηλαδή, και εδώ είναι και η μόνη μου διαφωνία. Το μόνο που το, το ζητούμενο δεν είναι να γίνουν δημόσια προσβάσιμε νέες πληροφορίες, αλλά το πώς θα γίνονται δημόσιες. Αντίστοιχη συζήτηση λοιπόν γίνεται και στην Επιτροπή εσωτερική αγορά και για τα high value data sets, δηλαδή τις, ε, τα σύνολα δεδομένων από ε, λεωφοριακές συνδέσεις, για παράδειγμα. Από αυτές όμως αφαιρούνται από, την, ε, από τις υποχρεώσεις για την δυνατότητα αναδόμησης ε, εγώ έχω μιλήσει με μια σειρά από εταιρείε, Google, Apple, Amazon. Μπορώ να ε, αγοράσω δεδομένο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ανασύσταση της ταυτότητάς μου. Δεν χρειάζομαι καν, αν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, τις δημόσιες πληροφορίες. Δηλαδή, γι' αυτό και θα ήθελα, ε, όταν συζητούμε τέτοια θέματα, να επιδεικνύετε την αντίστοιχη στάση και απέναντι στους ιδιωτικούς φορείς και όχι μόνο στις δημόσιες πληροφορίες. Ευχαριστώ. η Κομισιόν. Έχετε δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας για τα σχόλια. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχουν αλλαγές για τον πολιτιστικό τομέα στην πρότασή μας. Δεύτερον, πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι η οδηγία για την εκ νέου χρήση δημόσιων πληροφοριών πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό στις, στους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τις δημόσιες επιχειρήσεις, εδώ μιλάμε για κλάδους που έχουν σημαντικά σύνολα δεδομένων και ταυτόχρονα ε, έχουμε δει ότι υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα στην επαναχρησιμοποίηση αυτών των πληροφοριών. Γι' αυτό και εξετάσαμε πολύ προσεκτικά τον αντίκτυπο των μέτρων ε, που προτείνουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε υποβάλει μια πολύ ισορροπημένη πρόταση από αυτή την άποψη. Σχετικά με τις χρεώσεις, τα τέλη για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων ε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε οι μεγάλε εταιρείε έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να αγοράσουν μεγάλα σύνολα δεδομένων για 50-100.000 ευρώ, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσει εμποδίζονται. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε τις, το κόστο για τι δημόσιες πληροφορίε. Επίση, θέλω να κάνω και μια σύνδεση με μια άλλη πρόταση που έχουμε υποβάλει, την πρόταση για το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, το οποίο και συζητείται στο πλαίσιο του του νέου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και εκεί θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων που προβλέπει η οδηγία να εκτελούνται από την πλευρά των κρατών μελών. Για παράδειγμα, την, ε, το να καθίσταται δυνατά αυτά τα υψηλή αξία σύνολα δεδομένων ε, στο κοινό. Ευχαριστώ. Να δώσω λοιπόν ξανά το λόγο στον κύριο Ζαγοράκη. Εκτό από να ευχαριστήσω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ του συναδέλφου για τι πολύτιμε παρατηρήσει και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Παρά τι επιμέρους διαφορέ, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα υποστηριχθεί από σχεδόν όλε τι πολιτικέ ομάδε. Σα ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Σα ευχαριστούμε πολύ. Υπενθυμίζω 16 Οκτωβρίου, 2 το μεσημέρι, τροπολογίες. Τέλος. Λοιπόν, και με αυτό έχουμε ολοκληρώσει τη συνεδρίασή μας, εκτός από το ότι πρέπει να σας πω το τελευταίο. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου μεταξύ 7 το βράδυ και 8 και 45. Περίεργη μέρα, περίεργη ώρα. Ξαναλέω, 22 Οκτωβρίου, 7 με 9 παρατέταρτο στο Στρασβούργο. Επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Λοιπόν, ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για την παρουσία τους. Έχουμε και μια συνεδρία των συντονιστών. Τρεις, τέσσερις ε, συντονιστές βλέπω αυτή τη στιγμή. Κοιτάζω ε, και προς την Άλντε θα έρθει η Γιάννα Τούμ. Η Τερέζα θα έρθει. Ωραία, εντάξει. Θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και να ξανασυναντηθούμε εδώ σε 10 λεπτά, να κάνουμε μια μικρή βολτίτσα εδώ στο διάδρομο και συνεχίζουμε 5 και 5.